αποστολή και την επίσκεψη δηλαδή της υποεπιτροπής μας πέρσι. Θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ήθελα να σας επισημάνω ότι εκεί θα έχουμε και δημοτικές και εθνικές εκλογές σύντομα, και βουλευτικές δηλαδή, και βάσει της έκθεση της κυρία Ρώνα Σμιτ, της ειδικής ε, ε, για την Καμπότζη, θα δούμε κατά πόσον, μετά από όσα συζητήθηκαν στο Παρίσι, μπορούν να οργανωθούν αμερόληπτες αντικειμενικές και δικές εκλογές. Το Σύνταγμα, στο άρθρο 31, ε, τονίζει την σημασία που πρέπει να αποδοθεί στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς καμία διακριτική μεταχείριση οποιοδήποτε τύπο. Είναι πολλά τα παραδείγματα της εφαρμογής του νόμου με διακριτικές μεταχειρήσεις ή τέλος πάντων με ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο σε πολύ πολιτικοποιημένο κλίμα. Θα πρέπει λοιπόν η καμποτζερή νομοθεσία να εφαρμόζεται όντω και στην πραγματικότητα. Έχουμε εδώ τη χαρά να έχουμε την κυρία Γκάλερ τη Διεθνού Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να τη δώσω το λόγο για να ακούσουμε και τη δική τη άποψη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που καλέσατε την υπατερμοστία για να λάβει το λόγο σήμερα για την κατάσταση στην Καμπότζη. <clears throat> Θα ήθελα να φίξω διαφορετικά ζητήματα την κατάσταση των ε, υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις τοπικές εκλογές, τις καταπιέσεις ενδεχομένως και τις συγκρούσεις που παραμένουν ανεπίλητες. Τις προστριβές, σε κάθε περίπτωση. Η διαπίστωσή μας σήμερα είναι λίγο συγκεκριμένοι για την κατάσταση των ακτιβιστών. Πιέζονται, πιέζονται. Και δυσκολεύονται να φέρουν εις πέρας τη δουλειά τους. Και αυτό σε ένα τεταμένο προεκλογικό πλαίσιο. 26 ε, ακτιβιστές Αυτή τη στιγμή δέχονται πιέσει και είναι φυλακισμένοι, 17 είναι τη αντιπολίτευση. Για τι υποθέσει που αυτή τη στιγμή ε, βρίσκονται σε εξέλιξη, να σα αναφέρω την υπόθεση των ε, πέντε, όπω ονομάζεται, και τέσσερα μέλη τη μη κυβερνητική οργάνωση Ad Hoc, μια από τι μεγαλύτερε μη κυβερνητικέ οργανώσει και τι πιο γνωστέ στην Καμπότζη, και ένα μέλο τη ε, Εθνική Εφορευτική Επιτροπή που ήταν και πρώην μέλος της ad Αυτοί οι πέντε κρατούνται από τις 2 Μαΐου σε αυτόφορο εδώ και 9 μήνες για την άσκηση των καθηκόντων τους, για τη δουλειά τους, δηλαδή τη στήριξη, τη νομική και οικονομική στήριξη προς κάποιο μάρτυρα. Σε μια περίπτωση εξωσυγη... σύναψης εξωσυγικών σχέσεων όπου ενεπλάκη και ο κύριος Κεμσόκα, ο αντιπρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης. Πρόκειται για μια υπόθεση με ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη προβολή. Η ad hoc, η οργάνωση αυτή δέχεται ιδιαίτερε πιέσει. Νέα μέλη της ad πρόσφατα έχουν ε, προσαχθεί ο πρόεδρος του κόμματος της οργάνωσης έχει αυτοεξοριστεί γιατί φοβάται ότι μπορεί να δεχτεί πίεσης. Επίσης, ο νόμος του ε, συνασπίζεστε ε, πρόκειται να ε, εφαρμοστεί όταν ε, ολοκληρωθεί εκδίκαση των υποθέσεων, κυρίως η υπόθεση κατά της ad Βέβαια, ο νόμος που καταργεί το δικαίωμα του συνασπίζεστε, ε, ξέρουμε ότι αντίκειται στην διεθνή και τη σύμβαση του ΙΕ για την ελευθερία του συνασπίζεστε και έχει να κάνει με την πολιτική ουδετερότητα. Ε, η ad hoc θεωρείται ε, ότι από τον Νοέμβριο του 2017 με τα μέλη της κράτηση μιλάμε για μια κράτηση αυθαίρετη και ο ειδικό εκτετραμένο του ΟΗΕ, καθώ και τα μέλη του ΟΗΕ, έχουν καλέσει σε απελευθέρωση των ε, πέντε. Πάντως δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει η φάση αυτή της ε, και θα απελευθερωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Επίσης, ο Τεπ άλλη υπόθεση, ο οποίος φυλακίστηκε για τη συμμετοχή του σε μία πορεία, την Μαύρη Δευτέρα όπω ονομάστηκε, που καλούσε στην απελευθέρωση ακριβώ των πέντε όταν συνελήφθη δύο ακόμη ποινικά αδικήματα που είχαν παραγραφεί ε, ανασύρθηκαν εναντίον του. Το ένα είχε να κάνει με μια συμμετοχή ε, το 2013 σε άλλη πορεία, διαμαρτυρία, που ζητούσε την απελευθέρωση μιας ακτιβίστριας για την αρπαγή γεών, κατά της αρπαγής γεών. Είχε συλληφθεί τότε και εκείνη η ακτιβίστρια μια υπόθεση συμμετοχή δηλαδή σε ε, διαδήλωση το 2013 που μπορεί να οδηγήσει σε πενταετή κάθριξη. Άλλη υπόθεση, μας ενισχύει 10 Ιουλίου 2016, δολοφονήθηκε ένας σημαντικός πολιτικός ε, αναλυτής. Η δολοφονία αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο διαφανούς και αντικειμενή ποινικής δικαστικής έρευνας. Ως προς το προεκλογικό κλίμα, ακούσατε ότι διώχθησαν επανειλημμένος ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Κόμματος του ο Κέμ Σόκα, ε, βρέθηκε σε κατοίκον κράτηση για 6 μήνες και η Εφορευτική Επιτροπή για τις Εκλογές, η ΝΕΚ, καταγράφει 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους που δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν λόγω έλλειψης εγγραφής στις εκλογέ στους εκλογικούς καταλόγους. Επίσης, μέλη της ΝΕΚ που είναι και μέλη της αντιπολίτευσης ξαφνικά διώκονται και πάλι σήμερα γιατί ανασύρθηκαν παλιές ποινικές καταδίκες εναντίον τους. Όπως είπαμε, το δικαίωμα του ελεύθερου συνεταιρίζεστε ο νόμος αυτός έχει χρησιμοποιηθεί κατά της hoc, της ΛΙΝΚΑΓΚΟ και άλλων κυβερνητικών οργανώσεων στην ε, Καμπότζη. Επίσης, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχει περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης. Υπάρχουν και άλλοι νόμοι περιορισμού των ελευθεριών. Νόμος για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο και άλλη μία για την διαχείριση των γεών. Αυτά ε, πρόκειται να ε, ενεργοποιήσουν και πάλι την, ε, τις κτηματικές διαφορές. Το 2011 ήδη πολλές εκθέσεις κατήγγυλαν το σύστημα των εμπορικών προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κλάδο της ζάχαρης ιδίως προς την Καμπότση, στο βαθμό όπου αυτές οι εμπορικές προτιμήσεις έχουν εντείνει την ε, τάση αρπαγής γεών σε συγκεκριμένε περιφέρειες της χώρας ιδίω. Για τις υποθέσεις αυτές ενεργοποιήθηκε, ανέλαβε δράση μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώθηκε αυτό. Το Ευρωκοινοβούλιο όχι μόνο ενέκρινε αρκετά ψηφίσματα, αλλά και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξαν ιδιαίτερα δραστήριοι. Ε, το μορατόριο του 2012 ήταν καρπό του έργου του και δημιούργησαν μια ad επιτροπή που ανέλαβε να εξετάσει τις περιπτώσεις των θυμάτων αρπαγής γεών και να αποκατασταθεί η κάθε περίπτωση, δηλαδή να αποδοθούν και πάλι τα κτήματα στους ιδιοκτήτες τους. Σήμερα αυτά τα κτηματικά, αυτές οι κτηματικές ε, προστριβές, οι διαφορές δεν έχουν επιληθεί, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και οι ακροάσεις. Πρέπει όμως να γίνει αυτό για να λάβουν αποζημιώσεις τα θύματα και να ξαναπάρουν πίσω τα, δικαιώματά τους. τα δικαιώματά τους. Τα κτηματικά λοιπόν δεν έχουν επιληθεί. Το 2015 η Action Aid ε, ξέδωσε μία έκθεση για μια συγκεκριμένη περιφέρεια της χώρας. Το Μάιο του 2016 η πρώτη έκθεση παρακολούθησης για τη στρατηγική συνεργασία με την Καμπότζη τονίζει ότι οι αποζημιώσεις είναι ακόμη χαμηλότερε από αυτό που θα έπρεπε, το ότι είναι πάνω από 800 υποθέσει που δεν έχουν επιληθεί. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και η Γερμανία έχει ε, αποσυρθεί από τη χρηματοδότηση τη χώρα λόγω του θέματος των κτηματικών στην ε, Καμπότζη. Η Λίκαντο ε, μελέτησε πάνω από 70 νέε υποθέσει κτηματικών διαφορών με 9.000 οικογένειε να έχουν πληγεί. Και είναι εκατοντάδε υποθέσει στιματικών διαφορών που έχουν προκύψει και από τι αρχέ του 2016. Ο πληθυσμό θα πρέπει να μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του ε, και οι παραβιάσει αυτέ με τι αισθηματικέ διαφορέ να σοβούν. Μα ανησυχούν από τη στιγμή που υπήρξε μορατόριο για τι εμπορικέ προτιμήσει προ την Καμπότζη προστριβές ε, ξαναρχίζουν, γιατί οι εταιρείε αρχίζουν να εκμεταλλεύονται τα κτήματα της χώρας. Τις τέστε, στις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες το Plan Pen Post βλέπουμε τουλάχιστον έξι νέες περιπτώσεις κτηματικών διαφορών που έχουν να κάνουν με την ε, ζάχαρη. Τα καταγγέλει αυτά η Phnom Penh Post. Είναι πολλοί αυτοί που προσπαθούσαμε να τους ε, επιστρέψουμε τις, ε, τα κτήματά τους, αλλά ήδη από το Δεκέμβριο έχουν εκτοπιστεί και δεν μπορούν να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους. Μιλάμε λοιπόν για βίε συγκρούσει που οδηγούν σε απελπισία τον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει κανένα τρόπο να ε, λύσει το θέμα, το πρόβλημα. Να ολοκληρώσω με τρεις συστάσεις ενδεχομένως να ζητήσω από το Ευρωκοινοβούλιο να παρακολουθεί την κατάσταση προσεκτικά, ιδίω για τη δίκη του Τεκβανή, Τεκβάνη μάλλον, που θα λάβει χώρα στι 3 Φεβρουαρίου στι 2 το μεσημέρι. Επίση, να συνεχίσετε να ζητάτε την απελευθέρωση των 5, να υπάρξει έρευνα για την δολοφονία του Κενλή και ε, μια ε, μεταρρύθμιση των νόμων που έχουν πρόσφατα εγκριθεί. Επίσης θα ήθελα το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να καλεί την ΑΕΔ και την Γενική Διεύθυνση Trade να εγκαλέσουν, να απευθύνουν έκκληση προς την κυβέρνηση της Καμπότζης ώστε να τοποθετηθούν για το θέμα της επίλυσης των κλιματικών διαφορών και να δώσουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την ε, υλοποίηση και την εκπόνηση ελέγχων και κροάσεων για το θέμα των προβλημάτων στον κλάδο της ζάχαρης και των αδικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί στο πλαίσιο αυτό. Επίσης, το Ευρωκοινοβούλιο να καλέσει την ε, Γενική Διεύθυνση Trade, την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που διαθέτουν συμπεριλαμβανόμενης της, ε, της έρευνας για το κόστος τη πρωτοβουλία ε, τα πάντα εκτό από τα όπλα και για τι εμπορικέ προτιμήσει, εάν η κυβέρνηση τη Καμπότζη δεν ε, απαντήσει ικανοποιητικά στι συγκεκριμένε εκκλήσει που θα τι απευθυνθούν. Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λοχμπίλερ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι εξαντλητική η εικόνα που μας παρουσιάσατε και τοποθέτηση. Έχω ε, ερωτήσεις για την προετοιμασία ενώπιση των εκλογών. Είπατε ότι δεν έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους πολλοί πολίτες. Εξ όσων γνωρίζω, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διαπαιδαγωγήσει τους πολίτες και να τους κάνει να ψηφίζουν. Πώς γίνεται αυτό, για ποιο λόγο δεν έχουν εγγραφεί τόσοι πολλοί. Όταν πήγαμε στην Καμπότζη, ακούσαμε ότι πολλοί ε, εργάζονται στο εξωτερικό ως μετανάστες και δεν έχουν την ε, ευκαιρία ούτε τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Ε, πέρυσι μας είπαν ότι απέχει πάρα πολύ αυτό το ενδεχόμενο να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους οι εργαζόμενοι στο εξωτερικό. Εσείς τι λέτε, Πώς το αξιολογείτε, να πιέσουμε, υπάρχει ενδεχόμενο να περάσει, γιατί από ό,τι φαίνεται ε, ε, όσοι εργάζονται και ζουν ε, στο εξωτερικό αισθάνονται πιο ελεύθερα για να ψηφίσουν ελεύθερο εκείνο που θέλουν από εκείνους που ζουν στην Ήπεθρο. Τώρα, τι μεθόδους έχουμε εμείς και τι δυνατότητες να πιέσουμε την κυβέρνηση. Δεν αναφέρατε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να επιβάλλουμε μεμονωμένες ε, κυρώσεις, ατομικές δηλαδή, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά υψηλά ισταμένων προσώπων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που γίνει έρευνα σε βάθος ε, για την ε, δολοφονία του κυρίου Κέμλι που είναι ακτιβιστής και δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν με ηγέτης ενός μικρού κόμματος αντιπολίτευσης. Στις συζητήσεις που είχαμε με βουλευτές ε, της Καμπότζη, στην Πνομπέ, είπε, μας είπαν να το κοιτάξουμε και αυτό μήπως έχουμε στοχευμένες κυρώσεις ατομικά έτσι, εις βάρος κάποιων προσώπων. Επίσης, όταν πήγαμε εκεί, Είχαμε μακρές συνεδριάσεις με εκπροσώπους του δικαστηρίου που δικάζει τους κόκκινους χμέρ. Νομίζω δύο είναι οι δικαστικές αποφάσεις πρώην ηγετών των κόκκινων χμέρ και θα πρέπει να δικαστούν και άλλοι. Αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει να τους δικάσει ε, διότι λέει οι άνθρωποι αυτοί είναι ακόμα ενεργοί σε διάφορα πόστα και σε διάφορες θέσεις ε, δημόσιες στη χώρα. Για μια ερώτηση προς την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, άκουσα ότι Παράλληλα με την κηδεία κατά τη διάρκεια της κυρίας και του κυρίου Κεμλή διοργανώθηκε μια διαδήλωση κατά της καταστολής ε, ο κόσμος κατέβηκε φορώντας ε, ε, μαύρα μπλουζάκια. Και πολλοί έχουν φύγει στο εξωτερικό από αυτούς γιατί φοβούνται και ακτιβιστές. Και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το έχει ενθαρρύνει και το έχει υποστηρίξει πάρα πολύ. Και ε, πόσο χρησιμοποιείται η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να υποστηρίζει ε, η ad hoc για ε, ανθρωπίνα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Άλλο βουλευτή. θα δώσω στην υπηρεσία εξωτερικής Δράση το λόγο. Ο κ. Μάριο μπορεί να ξεκινήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να επαναλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει συνεχώς να υποστηρίζει την Καμπότζη στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Περίπου 7% είναι ο ρυθμός ανάπτυξης το έτος. Μεγάλη πρόοδος για τη μείωση της φτώχεια έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχεδόν διπλωσιάσει την αναπτυξιακή βοήθεια, περίπου 410 εκατομμύρια για 2014-2020 και επίση είναι μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά Ευρώπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2015 4 εκατομμυρια ευρώ ήταν εξαγωγέ Καμπότζη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρόσφατε ευρωπαϊκέ αγορέ στα προϊόντα εκτό όπλων ήταν κινητήρια δύναμη σημαντική για την ανάπτυξη στην οικονομική τη χώρα. Καλωσορίσαμε τα βήματα που έκανε η Καμπότζη όσον αφορά τι ανησυχίε των πολιτών για τι εκλογέ του 2013, ούτω ώστε να γίνουν μεταρρυθμίσει όσον αφορά την Εθνική Επιτροπή των Εκλογών, του καταλόγου των ψηφοφόρων και τι διαδικασίε εκλογικέ. Όμω, Παρά σημαντική πρόοδο παραμένουν πολλά προβλήματα. Το 2016 η Καμπότζη ήδη να αυξάνονται οι πολιτικές εντάσεις μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος, του CPP και, της, και του CNRP, της αντιπολίτευσης, με κρατήσεις και συλλήψεις μελών της αντιπολίτευσης, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και προσπιστών των οποίων δικαιωμάτων. Πιστεύουμε ότι τέτοιε δράσεις εν, εν ώψη των νέων εκλογών ε, δεν δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κατάλληλοι, ούτως ώστε όλα τα κόμματα και η κοινωνία των πολιτών να μπορούν ελεύθερα να παίξουν τους ρόλους τους. Ιδιαίτερα ανησυχούμε δε για τις παρατεταμένες κράτησης πέντε μελών της ΑΤΧΟΚ, ε, του οργανισμού του ΜΚΟ ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενός πρώην μελούς ε, και αποκαλούνται αυτοί οι κρατούμενοι οι πέντε του ad και ζήτησαν οι ειδικοί του ΟΗΕ την απελευθέρωση αυτών εχθές. Ο ειδικό της ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ επισκέφθη δύο φορέ την Καμπότζη το 2016. Εξέφρασε ανησυχίε για τον περιορισμό τη κοινωνία των πολιτών στην Καμπότζη. Και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενέβη του ΟΗΕ έχουμε κοινή δήλωση που εξεδόθη στι 14 Σεπτεμβρίου του έτου 2016 εκ μέρου 39 χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των 28 κρατών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, που εξάφρασαν πολύ μεγάλε ανησυχίε για την κλιμάκωση των πολιτικών εντάσεων στην Καμπότζη. Και δημιουργείται εντύπωση ότι είναι δυσανάλογη η νομική δράση που ασκείται κατά των επικριτών τη κυβερνήσεω. Μία δήλωση τη 20 Μαου του 2016 τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ζήτησε να σταματήσει η παρενόχληση δικαστική του ηγέτου τη αντιπολιτεύσεω και εκπροσώπων τη κοινωνία των πολιτών. Τώρα, σχετικά με τι επικείμενε εκλογέ, το 2017 και το 2018 έχουμε παρακολουθήσει πολύ στενά τη διαδικασία καταγραφής των ψηφοφόρων, κάτι που στήριξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία, η διαδικασία εγγραφής των ψηφοφόρων για τις ε, δημοτικές εκλογές του 2017 κατέληξε με 7,8 εκατομμύρια ψηφοφόρους, 81% του πληθυσμού που θα μπορούσε να ψηφίσει. Ετέθη ένα ερώτημα λοιπόν. Γιατί αυτός ο αριθμός δεν είναι υψηλότερος. Από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχουν πολλοί Καμποτζιανοί που ζουν στο εξωτερικό περίπου 1,5 εκατομμύριο οι οποίοι οι Καμποτζιανοί διανόμου δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει παράσχει υποστήριξη έδωσε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για εκλογικές μεταρρυθμίσεις εν ώψη των εκλογών του 2017 και του 2018. Θα συνεχίσουμε εμείς να στηρίζουμε τις εν λόγω εκλογές και θα εστιαστούμε επί της εκπαιδεύσεως και ενημέρωσης των ψηφοφόρων. Τώρα αυτές ε, οι διαμάχες όσον αφορά τα κτήματα ή την ιδιοκτησία της γης ε, συνεχίζεται στην Καμπότζη, συνεχίζουν τις επαφές με τις αρμόδιες φορείς, έκανε θετικά βήματα η κυβέρνηση Καμπότζης, όμως η πρόοδος είναι αργή όσον αφορά την επίλυση των διαφορών, όσον αφορά την ιδιοκτησία γης. Το έχουμε θέσει αυτό στην κυβέρνηση, θα πρέπει να δημιουργήσει φορέα ανεξάρτητο όσον αφορά τις διεκδικήσεις ε, γεών και διάφορα δικαιώματα που έχουν χωρηθεί για την καλλιέργεια ζάχαρης, φυτών που παράγουν ζάχαρη. Περιμένουμε ακόμα κάποια συγκεκριμένη κίνηση. Είναι μεγάλη προτεραιότητα για μας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εξακολουθούμε το θέτουμε στην κυβέρνηση. Ανησυχούμε τα μάλα για την όλη κατάσταση. Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Και σα διαβεβαιώνω ότι ο Επίτροπος Υπεύθυνο για το η κυρία Βάλστρομ, παρακολουθεί το θέμα εκ του σύνεγγης, πάρα πολύ προσεκτικά υπήρξαν θετικές εξελίξεις προς το τέλος του έτους 2016. Ε, δηλαδή, ο Κεμψόκα ε, ε, δεν απειλείται πλέον από σύλληψη. Δόθηκε αμνηστία βασιλική, δόθηκε χάρη. Συνεχίστηκε μία με μποϊκοτάς της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της υπηρεσίας της ΥΠΑ της εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα τελικά υπεγράφει, παρατείνεται μέσω μνημονίου, η παρατείνεται η παραμονή του γραφείου μας εκεί. Θα συνεχίσουμε να παροτρύνουμε την Καμπότζη να ενισχύει τη δημοκρατία και να δημιουργεί τις αναγκαίες συνθήκες για μια πραγματική διεξαγωγή των εκλογών με ένα δίκαιο σύστημα και έτσι τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι αποδεκτά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ε, πιστεύουμε πράγματι ότι είναι προς όφελος της Καμπότζης και για τη σταθερότητα της χώρας, τη μακροπρόθεσμη, θα ήταν χρήσιμο να διεξαχθούν εκλογές ε, που τη σε εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων και αυτό είναι δυνατόν μόνο αν μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερα η αντιπολίτευση και τα κόμματα αυτής, ε, χωρίς παρενόχληση και φόβο. Τώρα, όσον αφορά κάποια από τα τεθέντα ερωτήματα των Ευρωβουλευτών, στοχευμένες κυρώσεις. Αυτό θα πρέπει να επιβληθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για την ώρα δεν βλέπουμε ότι φύσταται κάτι τέτοιο. Πολύ σοβαρή επιδείνωση με άλλα λόγια της καταστάσεως θα οδηγούσε στην επιβολή αυτών των κυρώσεων. Τώρα στο θέμα των έκτακτων αυτοδικαστηρίων στην ε, Καμπότζη. 23 Νοεμβρίου του 2016 το ανώτατο δικαστήριο που επιβλέπει αυτά τα ειδικά δικαστήρια προέβλεψε ισόβιες ποινές για τον Κιώσαν Παν και την Ιωσέρ, ηγέτες των Ερυθρών Χμέρ, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όσον αφορά την εκένωση της Πνομπέχ αμέσως μετά την πτώση της πόλης στις 17 Απριλίου του 1975 εκδώσαμε μια δήλωση που υπογράμμιζε τη σημασία που έχει η απόφαση. Θεωρήσαμε ότι σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και όσον αφορά την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για σοβαρά, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά θα περιμέναμε το δικαστήριο αυτό να συνεχίσει το έργο του. Τώρα σχετικά με τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα συνεχίσουμε να θεωρούμε το θέμα είναι προτεραιότητα, έχει προτεραιότητα. Θέλουμε να εξετάζουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις και να τους υπερασπιζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που τα ανθρώπινα δικαιώματα στον βαθμό του δυνατού. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρέπει λίγο να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ο κύριος Χόσκιντς της Γενικής Διευθύνσεως ΔΕΦΚΟ έχει το λόγο. Τρία λεπτά, άντε τέσσερα σας δίνουμε. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι αρκετά σύντομος. Ο συνάδελφός μου της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης συνόψισε πολύ ξεκάθαρα το θέμα και τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις. Να επαναλάβω ότι όσον αφορά τις εκλογές έχουμε ένα πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων που υποστηρίζει την Εθνική Επιτροπή των Εκλογών για τη δημιουργία υποδομών και για καταχώρηση βιομετρικών στοιχείων και θέλουμε να την στηρίξουμε όσον αφορά την εκπαίδευση και την ενημέρωση των ψηφοφόρων και την, την να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών να επιτηρεί τις εκλογές. Αυτά υποστηρίζουμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή Διεξαγωγής των Εκλογών και οι σχετικές υποδομές θα είναι έτοιμες για να διεξαχθούν εκλογές στα πλαίσια ύψη των προδιαγραφών και θέλουμε να υπάρχει παρατήρηση πλευρά των κοινωνία των παρατηρητών, ε, κοινωνία των πολιτών, συγγνώμη. Και για τι δημοτικέ εκλογέ και τι εθνικέ εκλογέ να γίνουν σωστά και να ενημερωθούν καταλήλω οι ψηφοφόροι. Και θέλουμε ε, να υπάρχει παρατήρηση κατά τη διάρκεια τη εξογής των εκλογών και για τι δημοτικέ εκλογέ και για την Εθνοσυνέλευση. Τώρα, όπω είπε και ο συνάδελφο, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ που έχουν διατεθεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στηρίζουμε διάφορες στοιχείες αυτών. Στα πλαίσια στηρίξης δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστήριξης και της κοινωνίας των πολιτών και για το σχετικό πρόγραμμα για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκηση. Καλύπτουμε τι εκλογέ, δικαστικό κλάδο, προσπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επίλυση ε, προβλημάτων για την διοκτησία γη εμπόριο ανθρώπων, να ενισχύσουμε τη θέση τη γυναίκας στην κοινωνία. Λοιπόν, για το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για Δημοκρατία και Ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε 8,1 ε, εκατομμύρια για το 2016-2017. Θα χρησιμοποιήσουμε τη χρήση των κονδυλίων για την υποστήριξη διαφόρων τομέων που έχουν προτεραιότητα και κυρίως για την υπεράσπιση των προσπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέχρι τώρα έχουμε συνεργαστεί με αυτούς τους ανθρώπους για τα περιβαλλοντικά θέματα και τα θέματα διευθυνσίας γεών, αλλά οι ακριβείς προτεραιότητες ε, ε, για την πρόσκληση υποβολής ε, ενδιαφέροντος είναι κάτι που θα καθοριστεί στο εγγύ μέλλον συναρτής της καταστάσεως. Ευχαριστώ. Να σας δώσω και πάλι το λόγο. Πέντε λεπτά για να απαντήσετε στα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Για το θέμα των κυρώσεων Ναι, δεν έχουμε καταγράψει ακόμα τα χρηματικά ποσά των κυρώσεων που αφορούν τους διάφορους ε, σχετιζόμενους με αυτές τις ιστορίες αλλά θα την ε, έχουμε κατά την ιστορία αυτή. Επίσης να θυμίσω το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση από το 2012 και το πλαίσιο αυτό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιλύσει και να ασχοληθεί με προβλήματα που έχουν γίνει δυσεπίλητα. Τώρα, για το θέμα των κυρώσεων, να θυμίσω ότι η εισαγγελία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δέχτηκε προσφυγή για το θέμα αυτό ακριβώς της αρπαγής των γεών και τις πολιτικές συνέπειες αυτής της αυτών των περιστατικών που χαρακτηρίστηκαν ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητα. Λοιπόν, ε, ε, η τουλαχιστον αυτο ζητηθηκε θα υπαρχουν μια σειρα λοιπον απο νομικες που εχουν ενεργοποιηθει ηδη η καταπολεμηση της ατιμορρησία και το θέμα των κόκκινων πμέρων. Ήδη η Ομοσπονδία, η Διεθνούς Ομοσπονδία για τα Ανθρωπίνα Δικαιώματα έχει ασχοληθεί με το όλο το το Προεδρείο της Ομοσπονδίας στηρίζει το ψήφισμα για τις περιπτώσεις αυτές και συνεχίζει να μελετά την υπόθεση για τις διαδηλώσεις της Μαύρης Δευτέρας όπως ονομάστηκε η Ομοσπονδία και πάλι προσφέρει στήριξη για την κράτηση των υπερασπιστών των ανθρωπινών δικαιωμάτων και των ακτιβιστών σχεδιάζουμε συγκεκριμένε δράσεις και σε αυτό το πλαίσιο η Ομοσπονδία παρακολουθεί και την υπόθεση του ΤΕΠ Βάνη. Και όπως είπαμε και θα παρακολουθήσει και τη δίκη του στις 3 Φεβρουαρίου στι 2 το μεσημέρι. Νομίζω ότι κάλυψα τα συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν για την κατάσταση σε σχέση με τις εκλογές. Την παρακολουθούμε στενά με τα συγκεκριμένα με τα επιμέρους μέλη μας, την Λικάντο και την Ad hoc. Όπως είπα, το τοπίο είναι περίπλοκο, είναι δύσκολο και είναι σαφές ότι η κατάσταση καταστολής των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει να κάνει προφανώς και με, το με την προεκλογική περίοδο. Το θέμα των ε, γεών, των κτηματικών διαφορών δηλαδή, δεν μπορεί παρόλα αυτά να θαυτεί μέχρι να γίνουν οι εκλογές το 17 και το 18. Πρέπει να προχωρήσουμε και στα ντοσχέα αυτά αρκετά γρήγορα. Γι' αυτό χαίρομαι που άκουσα ότι παραμένει μεταξύ των προτεραιοτήτων για την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και διεξάγω το συμπέρασμα ότι θα υπάρξει έκκληση συγκεκριμένη προς την κυβέρνηση για να δούμε πώς προχωρεί η εξέταση του θέματος. Και ελπίζω να οργανωθούν σύντομα και σχετικές ακροάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πολύ για την προσέλευσή σας. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, κλείνοντας τη συζήτηση αυτή, είναι ότι ως ε, υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα παρακολουθούμε αδιάκοπα την όλη κατάσταση λόγω και των προθεσμιών των σημαντικών ραντεβού που μας περιμένουν οι δημοτικές και κοινοβουλευτικές εκλογές το 17 και 18 αντιστοίχως. Σας ευχαριστούμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για την Καμπότζη. Μετά θα περάσουμε στην Αγγόλα. Να ξεκινήσουμε Στην ημερήσια διάταξη έχουμε ενημέρωση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αγγόλα. Έχουμε μαζί μας τον Λουατή Μπεϊράου, ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μουσικό. Δεν ήθιστε να συναντούμε και να ακούμε ανθρώπους, πρόσωπα που υπάρχουν στα καταπήγοντα ψηφίσματά μας και συμπεριλαμβάνονται τα ονόματά τους. Σήμερα ο κύριος Εριράουα είναι γνωστός και στο χώρο της τέχνης ως ριζοσπαστικός ακραίος καλλιτέχνης, ερετικός καλλιτέχνης είναι από τους γνωστούς ε, καλλιτέχνες στην Αφρική και είναι γνωστός για τις καταγγελίες ε, που έχει κάνει κατά της κυβέρνηση της χώρας του για, την, ε, για το χειρισμό των εξετάσει το εισαγωγών πετρελαίου. Ο κ. Μπεράου έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα για τις δηλώσεις του αυτές και έχει πολλές φορές κρατηθεί κατοίκον. Είμαι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε λοιπόν μαζί μας και μπορούμε να σας ακούσουμε. Σας δίνω το λόγο. Σας ε, καλημερίζω θερμά κυρίες και κύριοι βουλευτές. Λέγομαι Λουάτι Μπεράου, είμαι πολίτης της Αγγόλας και της ε, Πορτογαλίας και ε, έχω εμπλακεί στην υπόθεση που ονομάζεται και 15 2 στην Αγγόλα. Σήμερα βρισκόμαι μπροστά σας ε, για να μιλήσω για το θέμα αυτό και ελπίζω ότι μπορώ να εκφράσω ε, την ε, θέση και των υπολείπων κατηγορουμένων στη δίκη αυτή για το ψήφισμά σας από τον Οκτώβριο του 2015. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμμετοχή της καθ' όλη τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης και με άλλες διπλωματικές πρωτοβουλίες που ήταν περισσότερο διακριτικές, αλλά το σύνολο όλων αυτών των ενεργειών άσκησαν πίεση στο απολυταρχικό καθεστώς της Λουάντα. Ε, αποφασίσαμε να αμφισβητήσουμε το από 41 χρόνια πολιτικό καθεστώς της Αγγόλας, ε, τα τελευταία χρόνια διότι δεχτήκαμε μέχρι και σωματικές επιθέσεις, ε, κάθε είδους, απειλές ε, κατά της ζωής μας, υπήρξαν ανεξήγητες εξαφανίσεις, δολοφονίες. Εδώ θυμώ τον, θυμούμε τον Ζαχαρίας Κασούλ και άλλους ε, διαδηλωτές που πλήρωσαν για τη ζωή τους, τη διαμαρτυρία τους. Το 2012 ήδη οι δολοφονίες ξεκινήσανε με δύο πυροβολισμούς, οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τη ζωή τους. Του πυροβόλησαν στο κεφάλι και του πέταξαν στους κροκόδηλου. Ο μηχανικό Ουμπέρτο Γκάντε από το 2013 έχει χάσει τη ζωή του. Το πυροβόλησαν στα πλευρά και το έγκλημά του ήταν ότι συμμετείχε σε μια διαδήλωση κλέβοντας πορτοφόλια ε, και όλα αυτά σε αντίθεση με τις δολοφονίες των δύο νέων κοντά σε μια περιοχή κοντά στο πρωταϊδικό Μέγαρο. Επίσης, ε, μία δημοσιογράφος από την Γουινέα έχασε τη ζωή της, χωρίς να μάθουμε ποτέ τίποτα πλέον για τα ίχνη της. Εδώ και ε, ένας μικρός με τον ίδιο τρόπο έχασε τη ζωή του. όταν προσπάθησε να εμποδίσει μια μπουλντόζα που θα κατεδάφιζε ένα κτίριο να περάσει, αλλά πλήρωσε και αυτός με τη ζωή του. Είναι πολλά τα θύματα λοιπόν της πολιτικής βίας και μέλη της αντιπολίτευσης, αλλά δεν χρειάζεται να τα πω όλα αυτά με λεπτομέρειες, γιατί νομίζω ότι τα γνωρίζετε καλά. Επίση, φαντάζομαι ότι δεν έχει καταφέρει να σα εξαπατήσει η κυβέρνηση τη Αγγόλας με την πολύ μέτρια ρητορική της το ψήφισμά σας αποδεικνύει ότι δεν έχει πετύχει εξαπάτηση. Θέλω απλώς να θυμίσω ότι 15 2 είναι μια δίκη που ε, κατηγορεί για ένα ανύπαρκτο έγκλημα. Η αμνηστία που δόθηκε είχε ανακαλέσει την ποινή που είχε επιβληθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Εμείς δεν θέλουμε καν αμνηστία. Θέλουμε από το Ανώτατο Δικαστήριο να ε, παραγράψει τελείως το υποτιθέμενο αδίκημα ή έγκλημα. Πρέπει να πούμε εδώ ότι τα θύματα έχουν ε, μετατραπεί σε κατηγορουμένους. Ο κύριος Σούμη, λόγω χάρη, έχει καταδικαστεί σε 28 χρόνια κάθεξης ενώ η νομοθεσία της Αγγόλας προβλέπει μέγιστη κάθριξη 25 χρόνια. Από τον Ιούλιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει με την Αγγόλα ένα έγγραφο που ονομάζεται Κοινή Υπορροία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αγγόλα και δεσμεύεται μεταξύ άλλων ε, μάτων υποσχέσεων η κυβέρνηση να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από τότε που συζητιούνται αυτές οι συμφωνίες ε, στη Λουάντα, δεν έγινε τίποτα αυτά με ε, μέλη του ΜΠΕΝΤΕ, του κόμματος της αντιπολίτευσης που διαμαρτύρονταν, να δέχονται επιθέσεις με σιδηρολοστούς. Επίσης, η εκπρόσωποι του κόμματος ε, της, ε, του κυβερνώντος κόμματος είχαν τουλάχιστον ένα λεπτό ε, τηλεοπτικού χρόνου ο καθένας για να μπορούν να υπερεφανευτούν για αυτό το φωτατόρθωμα. Το κοινοβούλιο ελέγχει το πώς κατευθύνονται τα διάφορα κονδύλια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο τελείως αυθαίρετο τα κονδύλια που καταβάλλετε εσείς και οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Θα ήθελα λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Πορτογαλία ιδιαίτερος, ώστε να ερευνηθεί η προέλευση του χρήματος που έρχεται από την Αγκόλα. Πώς ανοίγουν οι πόρτες για να ξεπληθεί το χρήμα αυτό στην Πορτογαλία. Είναι μια είσοδος, μια πόρτα για την Ευρώπη. Εσείς θα πρέπει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να απαιτήσετε η Πορτογαλία να συμμορφούνται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να μην δέχετε χρήματα τα οποία δεν είναι καθαρά. Η Αγγόλα ουδέποτε σκόπευε να τηρήσει κάποια από αυτέ τι συμφωνίε σε τι διεθνεί συμβάσει που κύρωσε. Δέχτηκε για ένα-δυο λόγου πολύ συγκεκριμένου. Ε, να παριστάνει ότι βρίσκεται στην πορεία του δημοκρατισμού ώστε να κερδίσει χρόνο και αξιοπιστία. Μέχρι να ε, κουραστούν χρόνο με το χρόνο με το χρόνο οι διάφοροι εταίροι και συνεργάτε να επιμένουν στι ίδιε απαιτήσει. Το 2017 είναι χρονιά εκλογών στην Αγκόλα, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Παρά τι δηλώσει των υπευθύνων για την εκλογική παρατήρηση από το 2008, 2011 και 2012, που θεώρησαν ότι σε γενικέ γραμμέ ήταν ελεύθερε και αμερόληπτε εκλογέ, οι εκθέσει δίνουν πολύ συγκεκριμένε λεπτομέρειε για τις βίες ενέργειες κατά τη διάρκεια του προεκλογικού ε, διαστήματος με την θύμωση ε, όλων των αντιφρονούντων και όσων διαφωνούν με το κυβερνών κόμμα. Με τη συνηθισμένη μας ε, υπεροψία βλέπουμε ότι πλέον δεν, δεν προβλέπονται παρατηρητές για τις εκλογές στην Αγγόλα. Κι όμω, η έλλειψη ανοχή σε πολιτικό επίπεδο, οι κρατήσεις κατοίκων, οι συνοπτικέ εκτελέσεις, οι δολοφονίε και οι διώξει, η καταπίεση των θεμελιωδών ελευθεριών παραμένουν ένα γεγονό. Θα πρέπει να πούμε ότι στη δική μας όρημη δημοκρατία ε, μπορούμε να παραλείψουμε τη δική σα αποστόλη παρατηρητών, Όμω, να είστε βέβαιοι ότι κάποιοι δημοκράτε, στο όνομα τη διαφάνεια, τη δημοκρατία και τη ανθρώπινη ελευθερία, κάποιοι ε, αμετανόητοι, ρισκάρουν ακόμα τη ζωή του. Επίση, η ΑΚΑΠ, ε, η γαλλική αυτή οργάνωση που δράστηκε στο Παρίσι και στι Βρυξέλλε, έχει διευκολύνει την ε, μάχη μα και χαίρομαι πολύ που επέτρεψε την οργάνωση αυτή τη συνάντηση. Οι βουλευτέ που βρισκόνται εδώ, η κυρία η και ιδίω οι κυρίε Αναγκόμε και Μαρίζα Ματίας. Εύχομαι να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την Αγκόλα, έστω και με γραπτά διαβήματα. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην Άννα Γκόμες, που ε, διευκόλυνε αυτή τη συνάντηση, από ό,τι ξέρω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη η χαρά που έχουμε μαζί μα τον Λουάρτι Μπεράου, που είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία όσων συζητούν για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, όχι μόνο στην Αγγόλα, στην γνωστό, αλλά και στην Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη. Ελπίζω να γίνει, γνωστή, να γίνει γνωστός ο αγώνας σε περισσότερο κόσμο στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό αυτό που μας, μόλις μας είπε ο κ. Μπεϊράου για τις σαφείς διασυνδέσεις μεταξύ των παραβιάσεων των δικαιωμάτων που διαπράττονται στην Αγγόλα και την διαφθορά. Την διαφθορά με κρατικούς ε, πόρους, ε, μάλιστα χρήμα κρατικό που μέσω του ευρωπαϊκού ε, χρηματοοικονομικού συστήματος ξεπλένεται στην Πορτογαλία. Γίνεται πλυντήριο της ε, Αγγόλας Πορτογαλία. Μα είπε ο Λουατή ότι κάποιοι ακριβώ αυτό προσπαθούμε να πολεμήσουμε και προσφάτω δέχτηκα επιστολή από την European Banking Authority, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, απάντηση που ε, είχε να κάνει με την δέουσα επιμέλεια η οποία ασκήθηκε για την παρακολούθηση των κρατών της Αφρικής και είχε να κάνει και με τη δράση του Πρόεδρου της χώρας και τις σχέσεις του με την ε, κρατική εταιρεία πετρελαίου, εκμετάλλευση των πετρελαίων πόρων της Αγγόλας εδώ διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των ευρωπαϊκών κανόνων για την καταπολέμηση του ξεπλήματος δρόμικου χρήματος και την ε, εφαρμογή τους. Φορείς όπως οι τράπεζες, και οι επιθεωρητέ των τραπεζών θα έπρεπε να έχουν να λάβει εδώ δράση και όχι μόνο. και επιχειρήσει εμπλέκονται και άλλοι. Θα ήθελα λοιπόν ο Λουάτη να μας πει ίσω περισσότερα, εάν ε, γνωρίζει, εάν μπορούμε να ξέρουμε περισσότερα στο Κοινοβούλιο για αυτό το ιερό τέρας ο οποίος έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. γιατί ακούγονται αριθμοί από 13 έως 30 έως 1.300 νεκρούς. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαστάσεις ε, της σφαγής αυτής. Ξέρω ότι η σφαγή υπήρξε πάντως και πολλοί έχασαν τη ζωή τους, ακόμα και γυναίκες και παιδιά. Επίσης, Ήθελα ο Λουάτη να μας πει ότι μπορεί, ότι γνωρίζει για το πώς βλέπει την κατάσταση αυτή τη στιγμή γιατί ένας ε, Πορτογάλος εισαγγελέας συνελήφθη ως συνένοχος σε προσπάθεια ο Μανουέλ Βισέντε, που είναι πρώην πρόεδρο τη Βουλή τη Αγγόλα και ε, μέλο τη αντιπολίτευση, να εμπλακεί σε δίκη εναντίον του. Θα γίνουν εκλογέ, δεν του δόθηκε το δικαίωμα να κατέβει στι εκλογέ, εφόσον ήταν κατηγορούμενο. Πώ τη βλέπετε αυτή την κατάσταση, Και επειδή ακριβώ θα γίνουν εκλογέ, Η ε, αρχηγοί τη αντιπολίτευση, ιδίω αυτό τη Ουνίτα και τη Κάζα, και στη Φιλαδέλφια, με παρουσία της κυρία Μογκερίνη και την ε, ε, διάσκεψη του κόμματο των Δημοκρατικών, εκεί συζητήθηκε για το αν πρέπει να υπάρξει αποστολή παρατηρητών στις εκλογέ φέτο. Όμως, η πληροφορία που έχω σήμερα είναι ότι δεν υπήρξε επίσημο αίτημα από την κυβέρνηση. Προφανώ κάθε κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει ευθύνη για να γίνονται σεβαστοί κανόνε ανεξαρτησία, ε, και δικαιοσύνης των ε, αποστολών παρατήρησης. Ξέρουμε ότι θα υπάρξει αντίσταση το 2012. Δυστυχώς τότε ο Ντουράο Μπαρόζο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε μόνος του ότι δεν χρειάζονταν ε, αποστολή παρατήρησης για τα νόριμη δημοκρατία η Αγγόλα. Ξέρουμε ότι διασυνδέσεις έχει ο Ντουράου Μπαρόζο με το καθεστώς της Αγκόλας και έτσι εξηγείται το πόρισμά του για τη μηγορία του. Όμω πρέπει κάπως να το πολεμήσουμε την αντίσταση της ε, κυβέρνησης κυβέρνηση τη για να ε, διεξαχθούν με τρόπο διαφανή και αντικειμενικό οι εκλογές Και βεβαίω να υπάρξει παρατήρηση ευρωπαϊκή και διεθνή του πώ ε, διεξάγονται αυτέ. Η κυρία Ματίας, ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε σχέση με αυτά που η Νομίζω ότι έθεσε ήδη αρκετέ ερωτήσει. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω τον ε, Λουάτι Μπεράου. Είναι σημαντικό εδώ να μιλήσουμε για ελευθερία και δημοκρατία και όχι μόνο για την Αγγόλα αλλά και την Πορτογαλία και ακόμη και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου λίγα ακούγονται για τα όσα συμβαίνουν στην Αγγόλα. Η βασική μου ανησυχία έχει να κάνει με την ε, διαφθορά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Κάποιοι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια λεπτομερέστερη έρευνα για το θέμα αυτό και βεβαίω δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν πρωτοσέλιδα στην Πορτογαλία με, με τον τίτλο «Τα μπός της Αγκόλα στην Πορτογαλία». Εγώ... Πρέπει να δεχτούμε ότι συνενοχή υπάρχει. Υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων ε, φορέων και οργάνων. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε και να εμβαθύνουμε. Να μάθουμε περισσότερα για την Αγκόλα, γιατί ο Μπαρόζο δεν είναι πια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε από τη Σκοπιά του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου να ε, επιδιώξουμε να καλύψουμε τα αιτήματα του Λουάτι Μπεϊράου δεν αρκεί η αδιαφορία και ούτε αρκεί ο παρεμβατισμό. Είναι η δική μα αρμοδιότητα να καταπολεμήσουμε την έλλειψη ελευθερία και είναι πολύ σημαντική η παρουσία σου εδώ. Ευχαριστούμε επίση για τη διοργάνωση αυτή τη ακρόαση, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και να συζητάμε το τι συμβαίνει στην Αγγόλα. Ευχαριστώ. Και τώρα, πριν σε δώσω το λόγο, Έχουμε τον κύριο Μπαρμπέντο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στο ψήφισμα που ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο. Ζητήσαμε από την αντιπροσωπεία στη Ρουάντα Λουάντα, μια υποχρέωση δέσμευση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μόνο ε, αυτό. Πού βρισκόμαστε όσον αυτό το θέμα. Μήπως σε μερικά λεπτά μπορείτε να μας ενημερώσετε, να κάνετε κάποιες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόεδρε, ε, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρακολουθεί εκ του ε, την κατάσταση των σχέσεών μας με την Αγγόλα. Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο. Η κατάσταση είναι κάτι που συζητήθηκε και παρατηρείται από την αντιπροσωπεία μας στη Λουάντα. Επίσης, έχουμε κοινό διάλογο που καλύπτει και τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Αγγόλα και όταν χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επενεύει με δημόσιες δηλώσεις. Ο διάλογος επίσης διεξάγεται και με την κοινωνία των πολιτών στην αντιπροσωπεία μας. Από την αντιπροσωπεία μας έχουμε επαφές με τους πολίτες ε, όποτε αυτό χρειάζεται είναι διαρκής και μόνιμη η δραστηριότητά μας για να παρακολουθούμε την κατάσταση εκεί με εκθέσεις που συντάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Βεβαίως ε, έχουμε επαφέ και με την κυβέρνηση, αλλά ε, και όχι μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για πάρα πολλά θέματα ε, κοινού ενδιαφέροντος Ευρώπης-Αγγόλας και ένα από αυτά τα θέματα είναι η περιφερική σταθερότητα. φυσικά όποτε ε, έχει να πει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικό επίπεδο με την Αγγόλα γίνεται, διεξάγεται αυτός ο διάλογος με το σωστό τρόπο, με συγκεκριμένη μορφή ε, θεσμική και σε καλό κλίμα. Θυμάμαι ιδιαίτερα ε, κάτι που είχε να κάνει με τη συμμετοχή της Αγγόλας στη διαδικασία Κίμπερλι και ήταν σημαντική στιγμή γιατί για πρώτη φορά έγιναν συζητήσεις εκεί σε σχέση με το σύστημα Kimberley που πρέπει να ανοίξει για την κοινωνία των πολιτών. Αυτή ήταν ε, μια πάγια απέτηση έτσι ώστε η κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει σε αυτό το διάλογο και μια άλλη σημαντική συζήτηση διεξέχθη το 2014, αν δεν απατώμε, ε, στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αναθεώρησή τους και τα βασικά σημεία που εθίγησαν τότε εκεί αφορούσαν την κατάρτιση ενός καταλόγου συγκεκριμένων ε, βελτιώσεων που ε, το και αυτά τα παρακολουθεί και τα ελέγχει όχι μόνο ο Οργανισμός Εθνών και εμείς. Και τα θέτουμε υπόψη των αρχών της χώρας. Και είναι μόνιμος και διαρκής ο διάλογος και η παρακολούθηση και στο παρελθόν και στο παρόν. Και η επαφή ε, είναι δεδομένη και διαρκής ε, και μόνιμος ο διάλογο σε τακτά χρονικά διαστήματα με την κοινωνία των πολιτών για να δούμε τι μπορεί να γίνει για να ενισχυθεί η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Με μικρόφωνο. Θέλω να πω κάτι για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, την τελευταία φορά που πήγα στην Αγγόλα ήμουν με την ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήγα ε, να επισκεφτώ ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον πρόγραμμα για την ενίσχυση των παιδιών των φαναριών, των παιδιών που ζουν στον δρόμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό project αυτό, ένα έργο το οποίο στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται χρήματα αυτό, γιατί το υποστηρίζαμε και αποσυρθήκαμε εκ τότε. Έχει ενισχυθεί η χρηματοδότηση και άλλη ερώτηση. Τι έχετε να μας πείτε για τις συζητήσεις που κάνετε με την κυβέρνηση της Αγγόλας σχετικά με την παρατήρηση των εκλογών ή δεν ασχολείστε καθόλου με αυτό το θέμα. Okay. Ε, για τις δύο ερωτήσεις που κάνατε, δεν μπορώ εγώ να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση για τη χρηματοδότηση. Αυτό αφορά περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και όχι την Υπηρεσία εξωτερική Δράσης. Για το δεύτερο αυτό που μπορώ να σας πω ε, συγκεκριμένα είναι ότι το ενδεχόμενο παρατήρηση εκλογών συζητήθηκε σε πολιτικό επίπεδο τον Νοέμβριο και είναι μόνιμη και διαρκή η προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθεί εκλογές και στην Αγγόλα και σε άλλες χώρες. Αλλά ε, αυτό το θέμα το θέτουμε παγίως, όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό φυσικά. Λέσλι Πήραν. Καλημέρα σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την πρώτη ερώτηση, για την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχω τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αυτό, το συγκεκριμένο έργο, αλλά θα το κοιτάξω και θα σας απαντήσω. Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω διαφόρων μέσων, ε, το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και με διάφορα άλλα μέσα, με διάφορα ταμεία για την ανάπτυξη. Το 2016 υποστηρίξαμε ε, με 7 εκατομμύρια ε, την κοινωνία των πολιτών ε, με ε, προκήρυξη για υποβολή προτάσεων εκδήλωση ενδιαφέροντος. Αυτά είναι τα κανονικά κανάλια για την εκπαίδευση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα παιδιών και γυναικών. Τώρα ε, στην εκλογική διαδικασία προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών για την παρακολούθηση της διαδικασίας και να εξασφαλίσουμε να έχουν πρόσβαση εκλογές και γυναίκες. Επίσης για την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη, για τις πιο ευάλωτες ομάδες πολιτών κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ε, και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάθε χρόνο είναι πάγια υποστήριξή μας και στην αντιπροσωπεία ε, στην Αγγόλα. Ε, θα ήθελα επ' ευκαιρία να σχολιάσω ε, την επιμονή και τις προσπάθειες των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ρισκάνουν τη ζωή τους για να βελτιώσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλω να ξέρω τη δράση τους αυτή γιατί είναι πολύ δύσκολες συνθήκες και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα. Συγγνώμη, η κυρία Ματίας, μία μικρή ερώτηση. Τη ΣΥΣΟ πώς την υποστηρίζετε όταν έχετε τόσα πολλά προβλήματα ε, να στηρίξετε ΜΚΟ στην Αγγόλα. Um, I mean, this is a very... Κοιτάξτε, ήδη το περιβάλλον στο οποίο κινούμεθα είναι πολύ περίπλοκο. Κινούμεθα και στο Μπαγκλαντές, στην Ερυθρέα. Βρίσκουμε εμεί τρόπους μέσω της οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να το στηρίζουμε κυρίως μέσω τη προσκλήση υποβολή ε, προτάσεων και ε, με, συνεργαζόμαστε με τι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για πρόσβαση στη δικαιοσύνη, νομική αρρωγή, να του αποφυλακίσουμε. Αυτό δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά έχουμε κινηθεί παρομοίω σε άλλε χώρε. Θέλω να δω τις λεπτομέρειες ότι κάναμε στην Αγγόλα, αλλά ε, υποστηρίζουμε τις οργανώσεις ε, κοινωνίας των πολιτών. Ο πρόεδρος μπορούμε Κυρία. Κυρία. Μπορούμε να έχουμε ένα γραπτό σημείο μας όσον αφορά τις ε, χρηματοδοτήσεις. Πρόεδρε, λέει κυρία Γκόμες, η γραπτή απάντηση να συμπεριλαμβάνει και δράση στον τομέα της ανάπτυξης. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσε ένα πρόγραμμα για τη διατροφή χιλιάδων παιδιών στην νότια περιοχή της χώρας που πέθαναν τα παιδιά από την πείνα και η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε καν. Χάρη στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σώσαμε τις ζωές κάποιων παιδιών. Μπορεί το σημείωμα να συμπεριλαμβάνει λεπτομέρειε για τα αναπτυξιακά προγράμματα, διότι μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα προγράμματα και για υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να συμπεριλαμβάνει. Ορίστε. Θα είμαι σύντομο Για τον ε, για το Μούντου Σούμι. Ούτε εμεί ξέρουμε ακριβώ τι συνέβη. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι ακόμη και σήμερα συνεχίζεται η, διο, η δίωξη αυτού του θρησκευτικού δόγματος και των μελών του τον ε, περσινό Αύγουστο μάθαμε ότι υπήρξαν και περισσότεροι ε, θάνατοι. Φτάσανε υποτίθεται τι εκατοντάδε, αλλά κανεί δεν μπορεί να επαληθεύσει τα στοιχεία. Ε, γιατί τον Μάιο του 2015, όταν έλαβαν χώρα τα γεγονότα, η κυβέρνηση έκλεισε με στρατιωτικά μέσα την περιοχή, την περιέφραξε και δεν μπορούσαν ούτε βουλευτέ να πάνε. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να, πάνε, να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για να δούμε ακριβώ τι συνέβη. Πολλά καταγράφηκαν, ε, διάφορε εκθέσει έχουν συνταχθεί, αλλά υπάρχει μια ε, προμελετημένη σιωπή που καλύπτει το θέμα και πολλοί είναι αυτοί που έχουν καλέσει την κυβέρνηση τη Αγκόλα. Μάλιστα, κάποιοι θέλουν να στείλουν και ανακριτική επιτροπή. Η κυβέρνηση απάντησε στεγνά όχι είναι θέμα εθνικής ε, κυριαρχίας, οπότε κάτι προφανώς υπάρχει που προσπαθούν να κρύψουν. Δεν ξέρουμε τι συνέβη, υπήρξε σίγουρα κάτι πολύ σοβαρό έγινε και ήταν, ε, είναι πολύ επικίνδυνη από ό,τι φαίνεται η κατάσταση με αυτό το θρησκευτικό δόγμα, το φως του κόσμου όπως ονομαζόταν. Επίσης για το σκάνδαλο της διαφθοράς δεν ξέρουμε ποιο πρέπει να αναλάβει. Ούτε η πορτογαλική δικαιοσύνη είναι τελείω αμερόληπτη και αντικειμενική. Ο τύπο με διαρκή δημοσιεύματα αφήνει να εννοηθεί ότι κάποια ε, πράγματα αποκρύπτονται, δεν έχουν υποθεί ανοιχτά όλα όσα συνέβησαν. Βέβαια υπάρχουν πολλά τα οποία παραγράφονται και μπαίνουν στο αρχείο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να ερευνούμε το όλο θέμα και να πιέζουμε την Πορτογαλία, γιατί εκεί είναι η κυρία είσοδο του βρώμικου χρήματο στην Ευρώπη. Ω προ του παρατηρητέ, το επίσημο αίτημα έχει φτάσει. Δεν ξέρω ποιε είναι οι προθεσμίε που πρέπει να τηρήσουν. Ε. Όλα έτσι κι αλλιώ είναι σε προετοιμασία, αλλά πρέπει να γίνει σωστή προετοιμασία. Εγώ δεν έχω τα συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά ελπίζω εντό τη ε, νόμιμε προθεσμίε να γίνουν όλα όπως πρέπει. Διότι όσοι δεν είναι μέλη της κυβέρνησης και δεν συμμετέχουν στο κυβερνών κόμμα θέλουν να υπάρξουν παρατηρητέ. Τώρα για την παρέμβαση, για τον παρεμβατισμό. Μέχρι πολύ πρόσφατα έχουμε χαρακτηριστεί τρομοκράτες Φαίνεται ότι εγώ έχω λάβει ριζοσπαστική εκπαίδευση για να κάνω τρομοκρατικές επιθέσεις όπως αυτές που έγιναν στο Παρίσι. Όλοι εδώ είμαστε τρομοκράτες στα μάτια της ε, κυβέρνησης της Αγγόλας. Και μπορούμε να έχουμε παρεμβατική δράση στην ε, κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία της Αγγόλας και την ελεύθερη άσκηση της δημοκρατίας. Τώρα για την ερώτηση του κυρίου, το οποίο δεν διατήρησε το όνομα, δεν κράτησε το όνομα, για τον συστηματικό και μόνιμο διάλογο με την ε, κυβέρνηση. Έρευνα υπήρξε. Υπήρξε μάλιστα ένα κονδύλι 7.000 δολάρια για να στηριχθεί η κοινωνία των πολιτών. Ξέρουμε πολύ λίγες οργανώσεις ε, ε, στη χώρα που να είναι και αξιόπιστες και πολλοί λίγε έχουν και την προβολή που πρέπει για τη δουλειά τους και την πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δικαίωμα στη στέγη, δικαίωμα στην προστασία που μπορούν να αποδεχτούν παιδιά τα οποία είναι θύματα εγκατάλειψη. Είναι ελάχιστε. Δεν θέλω να προσπαθήσω να απαντήσω κάτι που δεν γνωρίζω. Όμως, από το 2011 στο 2015, όταν συλληφθήκαμε, Είχαμε μόνο ειρηνικέ διαδηλώσει και πορείε στα πλαίσια τη νομιμότητα και όσων προβλέπει το Σύνταγμα τη Αγκόλα και ουδέποτε εγώ ή κάποιος από τους συναδέλφους που εμπλέκονται στην ίδια δίκη δεν ε, προσκληθήκαμε σε διάλογο με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι όμως έχουμε δεχτεί απειλές κατά της ζωής μα Έχουμε δεχτεί διώξεις και το μόνο που μπορούσαμε να δημοσιεύσουμε ήταν ε, μέσω του τύπου. Ε, αυτό που εμπλέκει, το γεγονός που εμπλέκει μια ευρωπαϊκή χώρα, όταν ε, βρέθηκαν δύο κιλά κοκαίνη στα, στις αποσκευές μου και οι αρχές της Αγγόλας έκαναν την επίσημη καταγγελία και απίφθηναν έκκληση προς τους πορτογαλικές αρχές να με συλλάβουν για την άφηξή μου στην Πορτογαλία. Εγώ αυτή τη στιγμή με τρόπο ε, αφαίρετο, αυτή τη στιγμή θα βρισκόμουν σε κράτηση. Απλώς έγινε αντιληπτό ευτυχώς ότι πρόκειτο για παγίδα. Κανείς δεν μας προσκάλεσε σε κανένα είδους διάλογο με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αγγόλα. Επισκέψεις έχουν υπάρξει από το 2015, σίγουρα ήταν τελευταία αυτή, ε, και ο πρέσβης της Πορτογαλίας ε, μετά την ε, πίεση από την κοινωνία των πολιτών της Πορτογαλίας και τις σχετικές με κυβερνητικές οργανώσεις μετά από μέρες και μέρες απεργίας πείνας μα συνάντησε αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να διοργανωθεί ένας διάλογος εσείς μιλήσατε και για την περιοχή της Αμαντίθα και την ε, ζώνη, την διαδικασία του Κίμπερλι. Και μιλήσατε για τα δαματορυχεία. Εδώ μιλάμε για μια ζώνη ιδιαίτερα στρατικοποιημένη ε, και παρουσία στρατού που εκτελεί όσους ε, παίρνουν, αναλαμβάνουν τον κίνδυνο και πάνε να ψάξουν ε, διαμάντια μόνοι τους, τους θύρες, Ακόμη και αστυνομικοί και στρατιώτες γενικώ ε, παρακολουθούν αυτή την περιοχή. Πάντως στην Καμπίντα οι εχθροπραξίες συνεχίζονται λένε ότι είναι περισσότεροι οι στρατιώτες από ότι οι πολίτες εκεί. Μιλάμε για δύο γεωγραφικές περιοχές, από τις πιο πλούσιες ε, σε πόρους, αλλά και τις πιο αδύναμες ως προς το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε στοιχεία από τις εκθέσεις που συντάσσονται, αλλά δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτές. Και αυτό δεν πρέπει να παραλείψω να το πω. Ευχαριστώ. Θα σας ευχαριστήσω που ήρθατε έχετε την πλήρη υποστήριξή μας για τη μάχη που δίνεται στην Αγγόλα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αρμοδιότητα δική μα σαν υποπιτροπή είναι να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο την προσοχή, να φροντίσουμε αυτά τα θέματα να εξετάζονται και να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να επομιστεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα το όλο θέμα, να επομιστεί περισσότερε ευθύνε. Ευχαριστώ. Έτσι εδώ ολοκληρώνουμε σήμερα αυτό έχουμε άλλο κομμάτι της συνεδριάσεως. Θα εκδώσουμε ανακοινωθέν τύπου όσον αφορά τις εκτελέσεις που επαναλήφθηκαν στο Κουβέιτ. Επτά άτομα εκτελέστηκαν, τέσσερις άντρες και τρεις γυναίκες. Θα εκδώσουμε ανακοινωθέν τύπου για το θέμα. Ευχαριστώ. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 6 Φεβρουαρίου.